Δεν. ναι. ότι Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας. Πρώτα μας να δώσω το λόγο στην κυρία Τσίμερ. Euh, κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να εκφράσω την σοβαρότατη ανησυχία μας μετά τη χθεσινή υιοθέτηση της Ουγγρική Βουλής και μάλιστα σπευσμένα μια σειρά τροπολογιών στο Σύνταγμα που μάλλον αντιβαίνουν στις θεμελιώδει αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο η ανησυχία εκφράστηκε και από το Συμβούλιο της Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκδηλη ανησυχία δείχνει και ο Ουγγρικό λαός θα ζητούσαμε από την αρμόδια ε, Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Δημοσίων Πολιτικών Ελευθεριών, να εξετάσει αμέσως τις τροποποίησεις αυτές του Ουγγρικού Συντάγματο, στα πλαίσια ε, της ε, έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πρακτικές ε, στην Ουγγαρία με βάση το ψήφισμα της 16 Φεβρουαρίου 2012. Επίση να δούμε και κατά πόσο είναι συμβατέ αυτέ οι τροπολογίε με, το, με την Επιτροπή με την ΕΣΤΑ και θα ήθελα να αναλάβουμε αμέσως πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, non era un point of order. Δεν ήταν διαδικαστικό όμως αυτό. Η κυρία Τσίμερ τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παραπέμψω και να επανέλθω στην έναρξη των εργασιών μας Εκτές, Εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι ε, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έκανε μία δήλωση με την οποία διαφωνούμε για την απέλευση τεσσάρων ευρωβουλευτών που συνελήφθησαν από το Μαροκινό στρατό στην ε, περιοχή του Σαχέλ. Ε, παρακαλώ να κάνετε διάβημα η Δυτική Σαχάρα. Να ελέγξετε παρακαλώ. Ήταν επίσημα την προσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μαρόκο και πρέπει να μεταβεί εκεί στη ζώνη Σαχέλ. E Ευχαριστώ. Θα ενημερώσουμε τον Πρόεδρο. Ο κύριος Βερχόφστατ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, πριν από λίγα λεπτά υπήρξε μια παρέμβαση σε σχέση με την κατάσταση στην Ουγγαρία. Είναι φανερό ότι, βάσει παρέμβασης, με τις τροπολογίες οι οποίες συνεκρίθησαν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο λαμβάνει η χώρα μια παραβίαση θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών. Η αίτησή μου προς εσάς, κυρία Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, είναι ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τεθεί στην ημερήσια διάταξη αύριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θα λάβει χώρα η συζήτηση μαζί με την Κομισιόν και με την Ιρλανδική Προεδρία. Γιατί το λέω αυτό γιατί το άρθρο 7 της συνθήκης, το άρθρο 7, επαναλαμβάνω, είναι απόλυτα σαφές. Το 1 τρίτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θέσουν το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί να το κάνει η Κομισιόν. Ίσως η ίδια κυρία Ρέντινγκ μπορεί να το κάνει. Γιατί έχετε τη δυνατότητα στη συνεδρίαση της Κομισιόν να προχωρήσετε σε μια διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 εναντίον της Ουγγαρίας ή αλλιώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κινητοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνεται είναι να τελειώσει αυτή η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στασβούργο χωρίς να υπάρξει μια να τελειωσει αυτη η συνοδος ολομελεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό της Ουγγαρίας και χωρίς κάποια δράση του Συμβουλίου ή της Κομισιόν. Και πράγματι, αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα είναι ότι ο κύριος Όρμπαν αυτή τη στιγμή μας περιγελά, μας κοροϊδεύει με τον τρόπο αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από το φίλο μου τον κύριο Ντόλ, ο οποίος έχει κάνει ήδη μια σειρά από για τα θέματα αυτά ένα μήνα πριν για τον κύριο Μπερλουσκόνη, θα ήθελα να του ζητήσω να έχει το θάρρος να σταματήσει το πολιτικό του κόμμα να υποστηρίζει τον κύριο Όρμπαν σε αυτή την κατάφορη παραβίαση των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτησή μου λοιπόν Συνεχίστε, συνεχίστε. Η αίτησή μου είναι να τεθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι σαφές το έτοιμά σας, ε, κύριε Βερχόφστατ. Ο κύριος Σάιερ, διαδικαστικό. Ευχαριστώ. Άκουσα τις ε, παρεμβάσεις των σοσιαλιστών, ε, δημοκρατών και φιλελευθέρων για την Ουγγαρία και Τη λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακούμε με μεγάλη σοβαρότητα ένα τον άλλον. Βλέπω όμω ότι οι φιλελεύθεροι και σοσιαλιστέ εθελοτυφλούν όταν έχουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρε που οι κυβερνήσει έχουν φιλελεύθερο ή σοσιαλιστικό συνασπισμό ή είναι κυβερνώντα κόμματα. Βλέπω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά δυστυχώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ουδέποτε δεν ακούσαμε τον κύριο Φερχόφστατ να καταδικάζει τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ρουμανίας όταν μπλόκαρε το συνταγματικό δικαστήριο και δεν μπόρεσε να δημοσιεύσει εκείνο την απόφασή του. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις είχαμε ε, την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εφαρμόζει διπλά μέτρα και σταθμά. Κάτι που, σημαίνει, που ε, σημαίνει ότι το θέμα της αναθεώρησης του Ουγγρικού Συντάγματος είναι ουγγρική υπόθεση, γιατί το άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης ε, επισημαίνει ότι το Εθνικό Σύνταγμα και οι συνταγματικές δομές μιας χώρας ανήκουν στην κυριαρχία της και αυτή είναι απαραβίαστη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις ε, θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές ε, της κοινή ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Αλλά σε ό,τι φορά την τέταρτη αναθεώρηση του, Ευρωπαϊκού Συντάγματο, του ε, Ουγγρικού Συντάγματος, ήδη το έχει καταθέσει στις διάφορες επιτροπές για αναθεώρηση, αλλά σε καμία προηγούμενη παρέμβαση δεν αναφέρθηκε τίποτα για, για την αναθεώρηση. Τι πρόβλημα έχετε με τη συγκεκριμένη τέταρτη αναθεώρηση του συντάγματος. Ποιο είναι το συγκεκριμένο ζήτημα που πιστεύετε τόσο πολύ πια παραβιάζει δεν είχατε πει τίποτα. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Τα πάντα παραβιάζει. Ναι, ωραία απάντηση. Ο κύριος Φερχόφστατ λέει ότι παραβιάζει τα πάντα αυτή η τέταρτη αναθεώρηση. Ναι, αλλά αφήστε τις γενικές απαντήσεις. Πείτε μας συγκεκριμένα. Πού εντοπίζετε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κράτους δικαίου στην τελευταία αυτή αναθεώρηση. Αν αποδείξτε το. Η Ουγγαρία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Κύριε Ζάιερ, παρακαλώ ολοκληρώστε, λέει η πρόεδρο. Ναι, θα τελειώσω. Αλλά θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι η Ουγγαρία πληρεί τι αρχέ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Και δεν έχει νόημα να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά και μεροληπτικέ διαδικασίε ει βάρο οποιασδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αλλιώ θα δημιουργήσουμε μια ένωση που αντί να ενώνεται διασπάται όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ. Στην ημερήσια διάταξη δεν προβλέπεται συζήτηση για την Ουγγαρία τώρα. Τελευταίο, λοιπόν στη συζήτηση αυτή, κύριο Σταβάρες. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω εισηγητή για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κράτου δικαίου και δημοκρατία στην Ουγγαρία, θα ήθελα να πω σε όλου του συναδέλφου ο κύριος Φερχόφστατ ε, μα παρέψει στο άρθρο 7, ο κύριο Άγερ στο 4, να σα παραπέμψω εγώ στο 2, που είναι η ουσιαστική ε, πρώτη αναφορά ε, στη συνθήκη και λέει ότι εδράζεται η Ένωση στα θεμελιώδη δικαιώματα, στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Και όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και τα θεσμικά όργανα έχουν άμεση ευθύνη να προστατεύουν και να προασπίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες αυτή η τροποποίηση του συντάγματο, η αναθεώρηση στην Ουγγαρία, θίγει αυτά τα θέματα από την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη εμπεραμβανομένων και των εξουσιών του Συνταγματικού Δικαστηρίου μέχρι την ελευθερία τη έκφραση. Στο πλαίσιο τη έκθεση για την Ουγγαρία, ήδη έχουμε τέσσερα έγγραφα εργασία και μεταξύ αυτών μαζί με το ΕΛΚ για την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη στην έκθεσή μας που θα έρθει για την Ουγγαρία θα επικεντρωθούμε και στην τέταρτη αναθεώρηση του συντάγματος και σε βάθος θα την αναλύσουμε. Στο μεταξύ καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στρέψει πλήρως τις προσπάθειές της και να επικεντρωθεί στο διάλογο της με την Ουγγαρία στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν δεν συζητηθεί αυτό το κείμενο, δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα που θα άξιζε να ασχοληθούμε με αυτό για την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ. Allora, prendo... Μάλιστα. Σημειώνω λοιπόν ότι υπάρχει πρόταση για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Θα παραπευθεί στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, που θα λάβει και τη σχετική απόφαση. Ας περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έκθεση Κορέρα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ.